Dámy a pánové, díky... Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, κύριε Αφού έγινε αυτή η ψηφοφορία, τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο τη μέρη δηλαδή το σημείο το οποίο αφορά την Ινδία και την εκτέλεση του Μοχάμετ Αφζάλ Γκούρου και τι συνεπιέ τη. Κύριο Σαρνέσκη, ο πρώτο συνάδελφο που έχει ζητήσει το λόγο και θα τον έχει για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από πέντε μήνες, το Δεκέμβριο, ήδη συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ο βασικός ε, κατηγορούμενος ήταν η πιο πολυπληθής ε, δημοκρατία του πλανήτη, η Ινδία. Νομίζω ότι σε αυτό το κοινοβούλιο έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συχνά δεν κατηγορούμε χώρες που συστηματικά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μάλιστα το κάνουμε τρόπο ιδιαίτερα βίαιο. Είναι πιο βολικό βέβαια να ξεχάσουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες και να επικεντρωθούμε σε άλλες περιοχές που είναι πιο δημοκρατικές από αυτές. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή την κατάσταση όταν κατηγορείται μια χώρα που είναι πολύ πιο δημοκρατική από μια σειρά από άλλες χώρες. Αναφέρομαι στην απόφαση μετά από μια πολύ έντονη τρομοκρατική επίθεση. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καταδικαστική απόφαση. Ας το υπενθυμίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ψήφισμα Φυσικά δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις συνέπειες αυτής της καταδικαστικής απόφασης, αλλά μπορούμε να προβλέψουμε τις συνέπειες του ψηφίσματος ε, στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο στρατηγικό εταίρο της, την Ινδία. Αυτός ο στρατηγικός εταίρος είναι στο εδόλιό μας μετά από ούτε καν 6 μήνες. Το Δημοκρατικό μας Κοινοβούλιο μοντέλο της δημοκρατίας για πολλές χώρες του πλανήτη, με τη σειρά του επιτίθεται στη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη. Προβάλλοντας ένα φοβερό παράδοξο έτσι. Μια χώρα που έχει δημοκρατία, ποικιλομορφία και ανεκτικότητα. Ινδία. Επομένω, η Ινδία θα μπορούσε να αναζητήσει ένα άλλο εταίρο. Όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση πια. Όταν το Πακιστάν, Φερρυπίν, μια γειτονική χώρα της Ινδίας, παρουσιάζει συστηματικά περιπτώσεις βασανιστήριων, συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμείς το ξεχνάμε και επικεντρωνόμαστε στην Ινδία. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής. Η κυρία Ντελή η εκτέλεση του Μοχαμάντ Αφζάλ Γκουρού έγινε στις 9 Φεβρουαρίου και είναι ένα σημάδι α, ανησυχητικό ε, μια στάση στην Ινδία για την επανεμφάνιση της θανατικής ποινή. Είναι η δεύτερη θανατική ποινή μετά από τρεις μήνες. Ενώ είχε σταματήσει η Ινδία επί 9, επί 9 χρόνια συγγνώμη, να εκτελεί. Ε, πηγαίνοντας αντίθετα στο ρεύμα που υπάρχει ε, στον πλανήτη, δηλαδή 140 χώρες, περίπου 2 τρίτα των χωρών του πλανήτη, κατήργησαν την ε, θανατική ποινή. 90% των χωρών δεν εφαρμόζουν αυτή την ποινή. Ο Μοχάμεντα Αυσάλ Κουρού καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το Δεκέμβριο του 2002 ε, με βάση ένα νόμο για την πρόληψη της, δημοκρα... τρομοκρατίας. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για την ε, δίκαιη δίκη του. Δεν επέλεξε τον δικηγόρο του, ούτε είχε δικηγόρο σε όλη τη διάρκεια της δίκης του. Οι δικές αρχές πριν από κάθε εκτέλεση συνήθως έδιναν πληροφορίες για την άρνηση της αίτησης χάριτος κτλ. Σε αυτή την περίπτωση όμως ε, προέβησαν στην εκτέλεση με κάθε μυστικότητα και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Με αυτό το ψήφισμα υπενθυμίζουμε ότι είμαστε κατά της αντικής ποινής σε κάθε περίπτωση, όποια και αν η φύση, όποιες και αν είναι οι συνθήκες ε, του εγκλήματος. Η, η αθωότητα ή η ενοχή του ατόμου. Γι' αυτό ζητούμε από το, το Ινδικό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ένα μόνιμο μορατόριο για την εσχάτη των ποινών με σκοπό να την καταργήσει εντελώς. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόρκολα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη για το γνώση ότι με υποστήριξαν οι συνάδελφοι σε σχέση με το είχα να προτείνω να μπει στη μεσαία διάταξη το θέμα τη εθνική καταδίκης στην Ινδία. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ε, στα πλαίσια αυτού του ψηφίσματο ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο πρόκειται να συνεχίσει να υποστηρίζει την κατάργηση τη θανατικής ποινή. Ο Μοχάμετ Αυσάλ Γκουρού εκτελέστηκε το 2011 για έγκλημα που το 2002. Η εκτέλεση δεν έγινε σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται διεθνώ. Ήταν αθώο, αλλά πρόκειται για μόνο μία από τι πολλέ προμήθειε περιπτώσει που έχουν ε, συμβεί στην Ινδία. Η Ινδία αποφάσισε να σταματήσει το πάγωμα των θανατικών καταδικών και εκτελέσεων τέλο πάντων ε, που είχαν γίνει για μια οκταετία. Έγινε μυστικά η εκτέλεση, δεν ενημερώθηκε η οικογένειά του. Πάντω πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πάρα πολύ θετικό το ότι τώρα για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό αναφέρεται η διαδικασία του Κασμίρ στο κείμενο του ψηφίσματός μας. Το Φεβρουάριο του 2013 ο κύριος Αυζάλ Γκουρού εκτελέστηκε ε, στο εσωτερικό των φυλακών μετά από μια απόφαση του Ινδικού Κοινοβουλίου. Επίσης ο πρόεδρος της Ινδίας ε, αρνήθηκε να του δώσει χάρη. Οι συγγενείς του επίσης δεν ενημερώθηκαν για την εκτέλεσή του, παρά μόνο εκ των υστέρων. Επίσης, σε 43 χώρες ε, εξακολουθούν να εφαρμόζουν την εσχάτη των ποινών, μεταξύ των οποίων και στην Ινδία και έχουν εκτελεστεί τα τελευταία χρόνια 679 άτομα. Πρέπει να εμποδίσουμε την, τις εκτελέσεις, θα πρέπει να ζητήσουμε να εφαρμοστεί η μορατόριμου στην θανατική ποινή θα υπάρχει το δικαίωμα στη ζωή και δεν πρέπει τον ε, 21ο αιώνα να εφαρμόσουμε τη θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, επόμενος, ο μιλήσει είναι ο μιλησει ο Μπαίνει για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, τα συλληπιτήριά μου προ την οικογένεια του εκλειπώντο. Είναι καλώ για το παράδειγμα το ότι δεν ενημερωθεί η οικογένεια για την επικείμενη εκτέλεση. έγινε εκτέλεση και στη συνέχεια παρά την εκστατεία που έγινε δεν δόθηκε σωρό στην οικογένεια του. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες ανέκαθεν ήμασταν κατά της θανατικής ποινή για όλη την υδρόγειο και υπό ιεσδήποτε συνθήκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση συμφωνεί με αυτή την θέση. Παρ' όλα αυτά όμω έχουμε ένα σωρό χώρε. Ακόμη, ιδίω στην Νοτιοανατολική Ασία, που δεν έχουν παγώσει ε, την εκτέλεση των θανατικών καταδικών. Και δεν πρόκειται μόνο για την Ινδία που έχουμε τη δεύτερη στη τέτοια περιπτώση, αλλά σταμάτησε το πάγωμα των εκτελέσεων και στο Πακιστάν πρόσφατα. Η Ινδία είναι η πιο μεγάλη δημοκρατία στον κόσμο, όπω προελέχθη, και επομένω θα έπρεπε αντί να είναι ουραγό, να είναι πρωταθλητή όσον αφορά το πάγωμα τη Ανατολική Ποινή ή την καταργήσή τη. Αλλά βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συνεχίζεται η νευτική διαδικασία συνεχιζεται η ενευτικη διαδικασια στο Κασμίρ παρά τα ε, σαν ανομαλίες που είχαμε στην γεννήθη ε, διαδικασία και έχουμε διάφορους που έχουν καταδικαστεί, βρίσκονται στη φυλακή και δεν πρόκειται μόνο για μέλη απόσχεσης του κινήματος, είναι και άλλοι. Οπότε αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε ένα προηγούμενο το οποίο ξεκινάει και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό ε, αποτελεί χειραγώγηση για τις επερχόμενες ειδικές εκλογές. Οπότε θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτοί που κρατούνται και πρόκειται να, ε, εκτελεστούν βρίσκονται εκεί λόγω των πολιτικών του προπηθήσεων. Η Λεβιάστον και οι συνεργάτε τη ε, θα πρέπει να πιέσουν στο γίνεται ώστε να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βερζιά για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2011 όταν παρουσίασε η Ινδία την υποψηφιότητά της στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, δεσμεύτηκε να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως ε, καταψήφιζε την, ε, το ψήφισμα του ΟΗΕ υπέρ του μορατόριου για την θανατική ποινή. Ε, υπάρχουν εκατοντάδες άτομα που είναι μελοθάνατοι εδώ και παραπάνω από 10 χρόνια πολλοί από αυτούς και κάθε χρόνο 130 άτομα ε, εκτελούνται. Ο ειδικό εκπρόσωπος του, 2000, του ΟΗΕ που πήγε το 2012 στην Ινδία ε, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυξάνονται οι καταδίκες σε θάνατο όχι μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα. Η εκτέλεση του Αυζάλ Γκουρού είναι πραγματικά παραδειγματική από αυτή την άποψη. Γιατί δεν είχε δίκαιη δίκη, Οι συγκατηγορούμενοι του βεβαίως ευτυχώς είχαν διαφορετική μεταχείριση. Η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε για την ε, επικείμενη εκτέλεσή του και δεν ε, δώσανε το σωρό του στην οικογένειά του. Ε, εξαιτίας της εκτέλεσής του έγιναν σημαντικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ με όπου τις κατέστηλαν οι αρχές με φοβερή βία. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι άξιο για τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. Δεν μπορεί να υπάρχουν ε, τέτοιες εξαιρέσεις. Είναι μια ποινή βάρβαρη που είναι απαράδεκτη τον 21ο αιώνα. Θα πρέπει οι ειδικές αρχές να το ξαναδούνε και θα πρέπει να συνταχθούν με το άλλο στρατόπεδο, όπως καν επί 8 χρόνια από το 2004 στο 2012. Ο κύριος ε, Πόσελτ για ένα λεπτό. Herr Κύριε Πρόεδρε, η Ινδία ε, σε αυτή την περίπτωση μας ενοχλεί για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι εμείς σε επίπεδο αρχής καταδικάζουμε την ε, θανατική ποινή, ακόμα και όταν πρόκειται και για καλούς εταίρους όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ινδία. Δεύτερον, ο τρόπος αυτός εκτέλεσης της θανατικής ποινή είναι αναξιοπρεπής για τη δημοκρατία. Μοιάζει περισσότερο με ποινή που επιβάλλεται σε δικτατορία. Και το τρίτο και σημαντικότερο, κάνουμε έκκληση στην Ινδία και το Πακιστάν επιτέλους ε, να επιδείξουν θάρρος ε, και διάθεση συμβιβασμού για ε, το περίπτωση του Κασμίρ. Μιλάμε για μια πιθανή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πυρηνικέ δυνάμει του κόσμου. Αυτό μπορεί να αποτελεί κίνδυνο και για την ειρήνη στην Ευρώπη. Κατόπιν τούτου, ω Ευρωπαίοι, πρέπει και εμεί να ασχοληθούμε με το πρόβλημα του Κασμίρ και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματο στην τόσο δύσκολη στρατηγική περιοχή. Επόμενη είναι η κυρία Σέντσεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η βοήθεια η δική μας αφορά την περίπτωση που συζητάμε. Πρόκειται για την επίθεση στο Κοινοβούλιο το 2001. Αυτή είναι η κατηγορία που απευθύνεται στον ε, Μοχάμπετ Αφσάλ Γκουρού ε, εκτελέστηκε πρόσφατα παρέμεινε 10 χρόνια στη φυλακή από τη στιγμή που απορρίφθηκε η αίτηση χάριτος που είχε υποβάλει εκτελέστηκε κρυφά. Η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων. Υπάρχουν περίπου 155 και άλλοι κρατούμενοι που περιμένουν την εκτέλεση της ε, θανατικής ποινής εις βάρος τους. Η δική μας πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθεί μορατόριο και επίσης ε, θέλουμε να καλέσουμε την Ινδία να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων. Επόμενο μιλήτρια, η κυρία Ογιουλάντ. Ευχαριστώ πολύ. Οι σχέσεις μας με την Ινδία έχουν εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει λοιπόν να ομολογήσουμε ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία έχει βελτιωθεί τα μάλα, αλλά παρόλα αυτά κρεμούν σημαντικά θέματα. Ε, υπάρχουν δημοτικοί δημοκρατικές αρχές ε, που σιγά σιγά παρισφρίουν στην κοινωνία. Η Ινδία δουλεύει σκληρά για να είναι ένα θετικό παράδειγμα σε αυτή την ασταθή περιοχή, την εύτραυστη περιοχή. Λυπούμεθα πάρα πολύ που η Ινδία αποφάσισε να αναστείλει το μορατόριο για τη θανατική ποινή που διήρκησε περίπου 8 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ένα βήμα που την απομακρύνει από τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τις ανθρώπινες αξίες που είναι ανεκτήμητες ε, και στη Δημοκρατική Ένωση προφανώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ εκφράζω τις σοβαρές μου ανησυχίες όσον αφορά την αμεροληψία του δικαστικού συστήματος στην Ινδία και ελπίζω η κυβέρνηση της Ινδίας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποδείξει το αντίθετο. Τέλος, θέλω να καλέσω την κυβέρνηση της Ινδίας ε, με τη μορφή κατεπήγοντος να μην εκτελεί στο μέλλον ε, τέτοιου είδου ε, παρεμφερείς ποινές. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Λόχπιλντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο ψήφισμα που έχουμε καταθέσει ζητάμε η θανατική ποινή να ε, μετατραπεί σε ποινή κράτηση του καθηγητή Σίντα Παμπουλάρ για τον οποίο ήδη το 2011 εγκρίναμε ε, ψήφισμα. Ο καθηγητής Σίν ε, αντιφρονών πήγε στη Γερμανία και ζήτησε άσυλο ε, αφού βέβαια η οικογένειά του εντωμεταξύ είχε βασανιστεί. Στη Γερμανία δεν του χορηγήθηκε άσυλο λόγω του ότι έτσι ισχυρίστηκαν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να εκδοθεί στην Ινδία. Στην Ινδία λοιπόν τον συνέλαβαν και έκτοτε βρίσκεται έγκλειστο στη φυλακή 10 χρόνια σε απομόνηση 22 ώρες την ημέρα σε ένα πολύ μικρό κελί. Η ψυχική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αργότερα τα γερμανικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι ήταν λάθος η απόφασή τους, ότι η ζωή του στην Ινδία πράγματι κινδυνεύει. Εκ των υστέρων λοιπόν κάνω έκκληση προς την Ινδική κυβέρνηση να αφήσει ελεύθερο τον καθηγητή ΣΥΝ ή τουλάχιστον να μην τον εκτελέσει όπως και όλους τους άλλους που βρίσκονται έγκλησες φυλακές και να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ποινή κράτηση. Στη Μαδρίτη το Παγκόσμιο Συνέδριο συνέδριο που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο αυτού του έτους θα αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι ώστε η Ινδία αλλά και οι άλλες χώρες οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή οι χώρες αυτές να αποδείξουν ότι είναι πρόθυμες να αναστείλουν την πολιτική τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ο ο κύριος Ρόσοβιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ο Μοχάμετ Αφχάς Γκούρου ε, καταδικάστηκε γιατί συμμετείχε στην τρομοκρατική επίθεση. Ε, σε εκείνη την επίθεση πέθαναν εννέα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Η περίπτωση του Λονδίνου μας δείχνει ότι διαδίδεται η τρομοκρατία, πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα. Θεωρώ ότι η ποινή ήταν ανάλογη με την πράξη που διεξήχθη στην Ινδία, που διέπραξε στην Ινδία. Ε, επίσης μην ξεχνάτε ότι η Ινδία είναι μόνη της σε μια περιοχή του πλανήτη που στηρίζουν τη δημοκρατία. Αυτό τον αγώνα κατά της δημοκρατίας ακόμα δεν τον έχουμε κερδίσει. Δέχεστε από τον κύριο Πόσελτ μια μπλε κάρτα. Παρακαλώ, κύριος Πόσελτ. Συνάδελφε, έχω να σας κάνω μία ερώτηση. Και εγώ είμαι κατά τις ε, τρομοκρατίες, αλλά είμαι εξίσου κατά της ε, θανατικής ποινή. Γνωρίζετε ότι ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος του 20ου και του 21ου αιώνα, ο Πολωνός Πάπας, ε, ο Ιωάννης ο ήταν σε επίπεδο αρχής κατά της θανατικής ποινή. Ναι, ευχαριστώ συνάδελφοι. Οι περισσότεροι Πολωνοί πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε μαλακοί απέναντι στους ανθρώπους που ενεργούν με ανθρώπινο τρόπο. Κύριε Δέχεστε μια άλλη μπλε κάρτα από έναν άλλο συνάδελφο. Παρακαλώ. Mike. Μικρόφωνο. Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, εσείς θεωρείτε ότι η θανατική ποινή θα πρέπει να εφαρμοστεί απέναντι στους τρομοκράτες, έτσι δεν είναι, αυτό μας λέτε. Α, και απέναντι και σε άλλους εγκληματίες, ε, οι οποίοι διαπράττουν να ε, ιδεχθεί εγκλήματα. Τι πιστεύετε τελικά. Είσαστε υπέρ της ανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, όταν έχουμε δολοφονίες, ε, βασανιστήρια, στον Κουαντάναμο περίπτωση, όλα αυτά είναι δικαιολογημένα, επειδή υποτίθεται ότι είναι τρομοκράτες αυτοί οι άνθρωποι. Τι λέτε. Απάντηση. Θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμόσετε θανατική ποινή όταν έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία λόγω των πράξεών τους δεν ε, φέρονται πια με απάνθρωπο τρόπο. Δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε καν ως ανθρώπους. Είναι υπάνθρωποι. Όταν σκοτώνουν αθώους, οι οποίοι δεν έχουν ε, διαπράξει κανένα αδίκημα, πρέπει να θανατώνονται. Αντίθετα, δεν μπορούμε βεβαίως να καταδικάζουμε σε θανατική ποινή αθώους. Προφανώς όχι. Ο επόμενος, ο κύριος Κλάς, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βλέπω ότι θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε εδώ από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν μιλούμε για την εκτέλεση εθνικής ποινής για τις τρίτες χώρες, για την Ινδία έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα την Ισλαμική τρομοκρατία και συμφωνώ με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να διαχειριστεί κάπω το ζήτημα στην Αγγλική Όμως, όμως και εμείς από την πλευρά μας να προσέχουμε και να μην θεωρούμε θύματα τους τρομοκράτες. Θύματα είναι αυτοί που έπεσαν που, που, που, κατά τον οποίο έγιναν οι τρομοκρατικές πράξεις αυτών των τρομοκρατών. γιατί η τρομοκράτες είναι αιτία πολλών θανάτων και πρέπει να προσέξουμε τι λέμε στο ψήφισμά μας γιατί ξέρετε ο Αφζαλ είναι υπέρ, ήταν υπέρ της θανατικής ποινής μόνο που ήθελε να επιβάλλεται σε αθώους μην το ξεχνάμε αυτό ο πρόεδρος ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Μακοβέη για ένα λεπτό Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. η εκτέλεση 7 χρόνια μετά την επιβολή της ε, και η ενκρυπτό ε, εκτέλεσή της ε, αυτό έτσι κι αλλιώς δεν ήταν νομότυπο παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του κατηγορούμενου υποτίθεται με βάση ένα δίκαιο περί τρομοκρατίας το οποίο όμως δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς προδιαγραφές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου αγωνιζόμαστε κατά της θανατικής ποινής. 1455 κράτη του κόσμου έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή ε, και νομίζω αυτό πρέπει να κάνει και η Ινδία. Η Ινδία λοιπόν καλείται να μην εκτελεί πλέον κανένα και να εισαγάγει πάρα αυτά ε, μορατόριο στην ε, θανατική ποινή και μάλιστα αυτό να το προβλέψει και στην νομοθεσία της. Ε, επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Παλέκης δεν είναι εδώ, κατόπιν τούτο ο κύριος Ομπεμάη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το βρίσκω λιγάκι περίεργο το γεγονός ότι σήμερα μιλάμε για, τις, ε, για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδία. Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ και εκεί δεν συζητάμε τίποτα. Άδικο αυτό. Όσον αφορά την εκτέλεση ε, θέλω να πω ότι έχω απόλυτη κατανόηση με τα θύματα όμως ε, η εκτέλεση του κυρίου Γκούρου με βάση κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις ε, φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αναταραχές στη γενέτειρά του ε, στο Κασμίρ που έτσι κι αλλιώ ε, είναι η περιοχή όπου αποσύρονται οι τρομοκράτες. Δεν θέλω να συστήσω τίποτα στην Ινδία, θέλω όμως απλά να πω ότι οι εκτελέσεις οι οποίες είναι με βάση τα ήθη έθιμα των Ινδουιστών, κατά πόσον αυτές οι εκτελέσεις δεν ε, οδηγούν σε περισσότερους μάρτυρες. Η Ινδία θα πρέπει να σκεφτεί κατά πόσον ε, θα πρέπει να αποκλιμακώσει την ένταση μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Πρέπει βεβαίως ε, και να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά δεινά, αλλά όχι σίγουρα με επιθετικές πράξεις. Ο Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα θέλω να πω κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς είναι το δεύτερο ψήφισμα για τη θανατική ποινή στην Ινδία, το οποίο συζητάμε κάτι διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Το πρώτο ψήφισμα αφορούσε την καταδίκη του Νταφίλντερ Μπανσίγκ, που το αίτημα χάριτός του απορρίφθηκε το Μάρτιο του 2013 και τώρα για δεύτερη φορά προσπαθούμε να στείλουμε ένα μήνυμα στις Συνδικές Αρχές. Θέλουμε να καταλάβουν την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θανατική ποινή και να, πιστεύ... να δουν ότι θεωρούμε πως η ποινή αυτή είναι απάνθρωπη και κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεύτερον, ο Αυσάλ Κουρού εκτελέστηκε μυστικά. Η διαδικασία αυτή δείχνει την, το πόσο έφραστη είναι η ενευτική διαδικασία στο Κασμίρ, σε μια περίοδο που η Ινδία προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους γειτονές της. Η, η αποσταθεροποίηση του Κασμίρ νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη λοιπόν να συνεργαστούν για να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο πρόβλημα. Ευχαριστώ και τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Χιούμπνερ είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ακόμα μια φορά είμαστε μάρτυρες ανησυχητικών γεγονότων, απουσία της ανεκτικότητας, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και συγκρούσεις και ταραχές στα σύνορα με το Πακιστάν. Η καταδίκη του Αφσάλ Κουρού, ο οποίος συνεργάστηκε στην επίθεση εναντίον του Ενδικού Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο του 2001, ε, προκάλεσε μια κλιμάκωση διαμαρτυριών που τροφοδοτείται από Ισλαμικούς κύκλους του Κασμίρ. Αυτή η κατάσταση δεν θα πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους αυτό που συμβαίνει στην Ινδία. Ε, θα πρέπει να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Ο πρόεδρος παρακαλεί την ομιλήτρια να μιλάει λίγο πιο αργά. Παρακαλώ, μιλήστε φυσιολογικά. Ο επόμενος ομιλητής. Είναι... Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πάνω από 20.000 οι οποίοι περιμένουν να εκτελεστούν σε όλο τον κόσμο μέσα στις φυλακές και πρόκειται για μια ποινή βάρβαροι, αναξιοπρεπή, ε, έτσι καταπατάει το δικαίωμα στη ζωή και πρόκειται εμπασχετός για κάτι το οποίο είναι ανέκλητο. Έχουμε πληροφορίες για το πόσο αμφίβολης ισχύως ήταν η καταδίκη και η δίκη του γκρού. Αφιζάλου θα πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή. Να μην επιβάλλεται υπό καμία συνθήκη. Είναι κάτι τελείω κατά των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, θα πρέπει έτσι να ρυθμίσουμε και τα τη εξωτερική μας πολιτική ως οργανωσή και η εξωτερική υπηρεσία για την προσωπία μας στην Ινδία όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιέσουν για την κατάργηση της θανατικής ποινής και σε διμερείς επαφές με την Ινδία. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο και τώρα ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μιγκάλσκι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα αυτή η περίπτωση να γίνει μια δικαιολογία για να επιτεθούμε στην Ινδία. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει το θέμα της θανατικής ε, ποινής. Για... Μετά από κάποιους μήνες, για δεύτερη φορά, καταδικάζουμε την Ινδία, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε κάπου και το θεσμικό τους ρόλο, τους αγώνες τους που κάνουν στην δύσκολη αυτή περιοχή του πλανήτη Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες με τις οποίες ε, λειτουργεί η Ινδία. Και αυτό το συγκλονιστικό δράμα του Αφζάλ Γκουρού δεν πρέπει να γίνει η δικαιολογία για να κατηγορούμε διάφορες χώρες. Νομίζω ότι ο καθένα έχει δρά με του ε, δικού του λόγου, μέσα στι δικέ του συνθήκε. Ο καθένα θα πρέπει να σεβαστεί τον άλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ινδία και αντίστροφα. Δέχεστε μία μπλε κάρτα. Βεβαίω. Κοιτάξτε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πια τη θανατική ποινή. Έχουμε αποφασίσει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν αναγνωρίζουμε τη θανατική ποινή. Δεν δεχόμαστε ε, την θανατική ποινή γιατί είναι μια βάρβαρη συνθή... Ε, κατάσταση η θανατική ποινή. Αυτό είναι όλο. Είναι η ερώτηση, η απάντηση. Εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Είμαι υπέρ της θανατικής ποινής. Ο κάθε ένας έχει το δικό του σύστημα. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ε, τη θανατική ποινή. Θεωρούν ότι είναι αποτελεσματικό σύστημα αποτροπής και, και ισχυρότατο αντικίνητρο για τη διάπραξη διαφόρων εγκλημάτων. Το, τώρα, το αν θα πρέπει να εφαρμόσει τη θανατική ποινή ή όχι γενικά είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Εσεί λέτε ότι είναι βάρβαρη η θανατική ποινή. Και όμως είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα για να αποτρέψουμε του τους Και γενικά απάνθρωπε συμπεριφορές και εγκλήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο επόμενο ομιλητής είναι ο κύριο Σάβαν. Η κυρία διορθώνει ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το κοινοβούλιο πρέπει να προστατεύει το δικαίωμα όλων για μια δίκαια δίκη οι περισσότεροι από εμά. Άλλωστε, είμαστε κάθετα κατά της θανατική ποινή. Και εδώ είχαμε κατηγορία τρομοκρατίας, αλλά θεωρούμε ότι η θανατική ποινή παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή και μάλιστα με τρόπο κατάφορο. Η εκτέλεση του κυρίου Γκουρού θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ελληνική διαδικασία στο Κασμίρ. Και μπορεί με αφορμή αυτή την καταδίκη να έχουμε κύμα βίας. Είχε παγώσει η Ινδία τις ε, καταδίκες, αλλά έχουν τους τελευταίους μήνες δύο θανατικές καταδίκες. Ε. Οπότε τώρα το πρόβλημα έχει ξανααναγκύψει μετά από 8 χρόνια. Βλέπετε που τα Ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Ταμπάργια. Ευχαριστώ. Η εκτέλεση του Μοχαμέντα Αυσάρ Γκουρού με απαγχωνισμό ε, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι μυστικών εκτελέσεων στην Ιδία και επανάληψη των ε, θανατικών ποινών στην χώρα αυτή. Πολλοί ομιλητέ και η κυρία Ντελή μίλησαν για αυτό το θέμα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν. Αλλά υπάρχουν σοβαρότατε αμφιβολίε για την δίκη δίκη του κυρίου Αυσαγκουρού. Δεν επέλεξε τον δικηγόρο του. Είχε έναν ανεπαρκή δικηγόρο, δεν είχε επαρκή πείρα, ήταν άπειρο κτλ. Η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε και αυτό ακούστηκε για την εκτέλεσή του. Η σωρό του δεν έχει επιστραφεί στην οικογένειά του για την κηδεία και την, ε, τις τελετές αυτές Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ λογικό αυτό το ψήφισμα να υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Το υποστηρίζουμε. Καλό θα ήταν να το υποστηρίξουμε όσο να τον περισσότεροι ε, ευρωβουλευτέ γίνεται πέρα από τι πολιτικέ μα διαφωνίε. Ο κύριο Ρόμεβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε κάτι ακαδημαϊκό, κάτι φιλοσοφικό, διότι η καταδική ποινή είναι μια ανέκλητη ποινή, η οποία παραδείγματο μα τη ζωή είναι κάτι το οποίο ε, το έχουν προσωγράψει στην διακήρυξη των δικαιωμάτων όλα τα κράτη-μέλη του ΙΕ. Επομένω, δεν είναι καθόλου προφανέ το να πούμε ότι μία ποινή για κάθε δικαιωμένο στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το ότι πάρα πολλοί φορεί των δικαιωμάτων έχουν ε, διατυπώσει πάρα πολλούς ε, πάρα για την καταδίκη αυτή όσον αφορά την, την, την υπεράσπιση όσον αφορά επίση το πώ αποσπάστηκε η ομολογία του από του αστυνομικού. Επίσης δεν ενημέρωσαν πριν την εκτέλεση την οικογένεια και επίσης δεν τους παρέδωσαν τη σωρά. Μπορούν να τον αποχαιρετήσουν. Όλα αυτά μας οδηγούν στο ότι θα πρέπει να είμαστε κάθετα αντίθεση στην Αντιπινή υπό συνθήκες. Η κατάργηση τη θανατική ποινή βοηθάει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, βοηθάει στο να παγιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, θέλετε ε, μια μπλε κάρτα, μια περώτηση από τον κύριο Μιγκάλ. Κύριε Μιγκάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ που δεχτήκατε τη δική μου την μπλε κάρτα. Έχετε δίκιο που λέτε ότι δεν υπάρχουν ε, αποδείξεις ε, για το ότι η ε, θανατική ποινή είναι αποτρεπτική. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποδείξουμε με εργαστηριακές δοκιμές, αλλά θα συμφωνήσετε απλά με τη λογική ότι μια μεγαλύτερη ποινή αποτρέπει περισσότερο από μια μικρότερη ποινή. Ίσως ε, η θανατική ε, ποινή να είναι λοιπόν αποτρεπτική. Εσείς τη δέχεστε αυτή τη λογική. Όχι, κοιτάξτε, εδώ το βασικό θέμα είναι ε, το κατά πόσο ένα μέτρο ε, μπορεί να είναι ανατρέψιμο, αναστρέψιμο ή όχι. Όμως ε, όταν ένα μέτρο δεν είναι αναστρέψιμο νομίζω από αυτό δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεύτερη μπλε κάρτα από την κυρία Μορβάη, θα τη δεχτείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς επικρίνατε ε, σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια ε, ποινικών ε, διαδικασιών και πιστεύω ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό να παραβιάζουν τα δικαιώματα του κατηγορούμενου. Επίσης επικρίνεται την παραβίαση, την ισοπαίδωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά αυτά και τα δύο τα, έχουν κάνει οι Ηνωμένε Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά η δική σας η ομάδα, οι πράσινοι που εκπροσωπούνται από τον κύριο Ταβάρες έγραψαν μια κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουγγαρία και θέλουν την έκθεση αυτή να τη στείλουν στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μα πώς είναι δυνατόν να τα συνδυάζετε αυτά τα δύο. Πώς μπορείτε να εκπροσωπείτε και τις ε, δύο απόψεις. Ε, λυπάμαι, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό που λέτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε. Τι να πω, δεν λέω τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ και τελευταία ομιλήτρια, η κυρία Κρετού. Πρόεδρε, για Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι για πρώτη φορά που συζητούμε το ότι θα πρέπει να καταργηθεί η θενατική ποινή στην Ινδία αλλά και σε άλλες 40 χώρες πρόκειται μια προσπάθεια που θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε διότι η θανατική ποινή παραβιάζει ε, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα κυρίως στη ζωή δεν είναι αποτρεπτική περισσότερο από άλλες κυρώσεις όσον αφορά τη διάπραξη εγκλημάτων. 50 τόσες χώρες έχουν ε, καταργήσει τη θανατική ποινή. Άρα με την ευκαιρία τη καταδική του Αουζαλγκούρου θα πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπαθίε μας για πίεση προ την Ινδία. Ας ευθυγραμμιστεί η χώρα με τα διεθνή πρότυπα. Τότε θα απολαύσει της δικής μας, του δικού μας σεβασμού και εκτιμήσει. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Μια τέτοια χώρα με τέτοια παράδοση να έχει τόσους ε, χιλιάδες φυλακισμένους οι οποίοι να περιμένουν θανατική ποινία. Α στήσουμε τι προσχέσει του ΣΥΝΔΕ να καταργήσουν τη δυνατική ποινή. Ο πρόεδρο. Κύριε Έτιγκερ, κύριε Επίτροπε, τι τελικέ παρατηρήσει. Κυρίε και κύριοι, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας όσον αφορά την ε, εκτέλεση ε, του κυρίου Γκουρού στην Ινδία σε 9 ε, Μαΐου η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάθη Άστον, αμέσως μετά στις 11 Φεβρουαρίου ε, έκανε μια σχετική δήλωση και ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να καταδικάσει ή να, ε, να ε, αναστείλει την θανατική να πείσει άλλα κράτη να αναστείλουν τη θανατική ποινή. Αυτή λοιπόν η απόφαση και η εκτέλεση της ε, ποινή, αυτή ήταν η δεύτερη μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια όπου δεν είχαν εκτελεστεί θανατικές ποινές στην Ινδία. Η μία περίπτωση ήταν ο Καζάπ, ο οποίος ε, ήταν ε, ε, ο μόνος που επιβίωσε, στην επίθεση στο Μουμπάι. Και τότε λοιπόν εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για το ότι άρχισαν και πάλι να εκτελούνται θανατικές ποινές μετά από ένα διάλειμμα 8 ετών. Ο πρόεδρος της Ινδίας τις ε, τελευταίες εβδομάδες απέριψε μία σειρά ετοιμάτων χάριτος και ε, φοβούμαστε ότι θα επανέλθει η θανατική ποινή. Ε, βεβαίως υπάρχουν ε, περιπτώσεις που είναι κοντά σε τρομοκράτες, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν φυλακισμένοι για περιπτώσεις βίας, βιασμών. Ορισμένοι εξ αυτών έγιναν γνωστοί στην ευρύτερη δημοσιότητα και έχουν θίξει το θέμα αυτό και Ευρωπαίοι Ευρωβουλευτές παν Σιμπουλάρ. Θα θυμάστε την περίπτωση αυτή που μας ανησυχεί. Η απόφαση εις βάρος του έχει εκδοθεί πριν από 10 χρόνια, έχει απορριφθεί η αίτηση χάρτης που έχει υποβάλει και γι' αυτό το λόγο υποφέρει πάρα πολύ και η υγεία του. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι στην κοινωνία των πολιτών δεν επικρατεί σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια ε, με τα οποία ο πρόεδρος της Ινδίας ε, εγκρίνει αιτήσει χάριτος και με ποια όχι. Και γι' αυτό το λόγο ε, ανησυχούμε. Εμείς στηρίζουμε την Ινδία στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας και επίσης έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε το θέμα αυτό με το Δελχή. Ο αγώνας κατά της ε, τρομοκρατίας Πρέπει βέβαια να γίνεται, ε, ενώ παράλληλα γίνονται απόλυτα σεβαστά, ε, σεβαστές οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι η θανατική ποινή δεν είναι αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή δολοφονικών πράξεων ή ε, τρομοκρατικών ενεργειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ανταλλάσσει απόψεις με την Ινδική κυβέρνηση για τη θανατική ποινή, για την εκτέλεσή της. Το έχει πράξει αυτό στο παρελθόν και θα το πράξει και στο μέλλον. Κατόπιν τούτου πρέπει να προάγουμε τον ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει ξεκινήσει γιατί θεωρούμε ότι και ελπίζουμε η Ινδική κυβέρνηση σύντομα να μας ε, προσφέρει μια νέα προθεσμία έτσι ώστε ο διάλογος αυτός που πολύ συχνά έχει αναβληθεί επιτέλους να συνεχιστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας.